οι διορισμοί θα εγγραφούν, στα, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδριάσεων. Αν, υπάρχει, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις συνεπώς μέχρι τη στιγμή ε, που γίνουν δεκτά τα πρακτικά, οι προτάσεις